και αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις θεωρούμε ότι ισχύουν αυτά τα αιτήματα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 μαζί με τον πρόεδρο του, του Συμβουλίου θα ε, υπογράψω δύο πράξεις που ε, εγκρίθηκαν σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία και οι οποίες θα δημοσιευτούν. Δύο γραπτές δηλώσεις.